Good afternoon, dear colleagues. Γεια σας αγαπητοί συνάδελφοι, λέει ο Πρόεδρος. Καθίστε παρακαλώ, ούτως ώστε να μπορέσουμε ταχαίως να προχωρήσουμε. Έναρξη της καταστατικής μας συνεδριάσεως της συγκρότησης σε σώμα και τώρα ο σκοπός μας είναι λοιπόν να συγκροτηθούμε εις σώμα και να ε, εκλέξουμε πρόεδρο και τέσσερις αντιπροέδρου, όπως ε, ε, προβλέπει η διάταξη παριθμών 191 του κανονισμού του Κοινοβουλίου. Τώρα, η σειρά της εκλογής θα έχει ω εξή. Πρώτα ο πρόεδρος και κατόπιν και όπως ήδη είπαν ε, ε, όπως είπαμε έχουμε τώρα την, την, ε, την, απαρτία, τους 50, τους 15 συγγνώμη που απαιτούνται, οπότε ευθύς αμέσως τώρα παρακαλώ να μα υποβάλλετε τις υποψηφιότητες για την Προεδρία. Έχετε το λόγο. Και εμείς, λέει η κυρία προτείνουμε τον Λόπες Αγγιλάρ ως Πρόεδρο. Και τώρα, κύριε Λόπες Αγγιλάρ, δέχεστε. Okay. Εκτός μικροφώνου, γνέφει καταφατικά ο κύριος Λόπες Αγγιλάρ. Και τώρα, υπάρχει έτερος. Όχι, από ό,τι φαίνεται. Ε, και για αυτό και σας προτείνω να ψηφίσουμε διαβοής για τον Πρόεδρό μας. Congratulations. Συγχαρητήρια, λοιπόν, Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ, ελάτε και να καταλάβετε την αίθουσα του Προεδρείου και να προεδρεύσετε. the only point today. This is the only point. Consider the elections. And that will be it. And then the vice. Now we elect the vice chair. Okay, just let me express gratitude and then we proceed. Okay. Good afternoon, honorable members. Let me start by saying that I am... Αγαπητοί συνάδελφοι, γεια σα. Πρέπει να σα πω πρώτα πρώτα ότι με μεγάλη τιμή θα προεδρεύσω τη Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, διότι όταν ξεκινήσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόκειται για την πρώτη μου θέση την οποία κατέλαβα, στην οποία εξελέγει και οπότε γι' αυτό θα ήθελα να σα πω ειλικρινώ ότι ε, ήρθα εδώ ω καθηγητή Ευρωπαϊκού και Συνταγματικού Δικαίου και έχοντας αυτή την τιμή τον να έχω υπηρετήσει την χώρα μου, την Ισπανία ως Υπουργός Δικαιοσύνης, Επομένως, ως μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου της κυβέρνησης της χώρας μου, είχα την εντύπωση ότι κάτι ξέρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο, όμως έσφαλα. Έσφαλα. Οπότε, απλώς θα σας αναφέρω με ειλικρίνεια ότι έμαθα περί τίνος πρόκειται εις αυτά τα δυόμιση χρόνια. Και επομένως είναι μεγάλη μου τιμή τόσο ώστε να μπορώ να μοιραστώ αυτές τις εμπειρίε, τις δημιουργικές, με εσάς, τα μέλη της Επιτροπής των Ελευθεριών. Ταυτοχρόνως σας είμαι ευγνώμων δεν μπορώ παρά να σα ευχαριστώ την ευγνωμοσύνη μου, τι ευχαριστίε μου για την κατανόησή σα, διότι πολλέ φορέ ε, την κατανόηση δίνεται και επίγεια. Επίγεια. διότι έχουμε εδώ διάφορα συμβάντα, διάφορε εντάσει, διάφορα επεισόδια τα οποία θα πρέπει να περάσουμε ούτω ώστε να μπορέσουμε να διεκπαιρεώσουμε την σαρπαστική μα ημέρη σε διάταξη που θα πρέπει και οφείλουμε να συζητήσουμε κατά αυτήν την θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και θα με δω και. Κόντρα σε όλα τα προγνωστικά τελικά τέθησε σκίση η συνθήκη Και επομένω ο τομέα τη ε, ελευθερία, τη δικαιοσύνη κλπ. Ε, Επιτέλου ε, υπάρχει τώρα. Είχαμε πει στο προγραμματάκι για, για, για την Στοχόλμη κατά την Ισπανική Προεδρία. Στη συνέχεια δε είχαμε πάρα πολλή δουλειά μπροστά μας και είμαι βέβαιος ότι θα συμφωνείτε ότι πρόκειτο για κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ χρονοβόρο αλλά και πάρα πολύ προκλητικό. Και βεβαίως όμως ήταν επίσης και πάρα πολύ θετικό διότι μπορούσαμε να δουλέψουμε αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτή την Επιτροπή. Μία από τις πλέον, η πιο, η πιο, πιο δραστηρία στο Κοινοβούλιο ήταν η Επιτροπή μας. Διότι Έχουμε την περισσότερη ύλη από όλου. Οπότε και γι' αυτό και είμαι υπερήφανο που έχω την ευκαιρία να μπορέσω να βελτιώσω την κατάσταση με τη δική σα βοήθεια και κατανόηση και επομένω να μπορέσω να συνεργαστώ με εσά. οπότε και έχουμε όλα αυτά τα, τα ενδιαφέροντα κατά αυτού τους ε, προηγουμένους ε, μήνες ε, του θέματα του ασύλου, της μετανάστευσης, της σχετικής συνεργασίας, όλα αυτά τα θέματα τα προωθήσαμε κατά την Πολωνική Προεδρία. Και προσπαθήσαμε επομένω να κάνουμε ό,τι καλύτερο περνούσε από τα χέρια μας ε, και κατά την τρέχουσα Δανέζικα και κατά την επομένη την Κυπριακή, οπότε και θεωρώ ότι πρόκειται να τα περάσουμε πάρα πολύ καλά μαζί κατά αυτήν την περίοδο. Και πάλι σας ευχαριστώ ειλικρινά για την εμπιστοσύνη την οποία επιδείξατε εις το πρόσωπό μου. Και επομένως μου δώσατε την ευκαιρία να συνεχίσω την Προεδρία της Επιτροπής μας με όλες μου τις δυνάμεις. Με λίγα λόγια, σας ευχαριστώ. Proceed now to the election of the vice chairs. Και ευθύ αμέσω τώρα θα προχωρήσουμε στην εκλογή των αντιπροέδρων τη Επιτροπή των Πολιτικών Ελευθεριών. Οπότε και ευθύ αμέσω πρόκειται να ψηφίσουμε για την ε, ε, εκλογή μέχρι και τεσσάρων ε, αντιπροέδρων. Οπότε παρακαλώ τώρα υποβάλλετε και χωρισμένα τις προσφυγιότητες ε, για κάθε ε, θέση. Ε, πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο. Κατόπιν δε θα ζητήσουμε από τους ενδεχόμενου υποψηφίου να αποδειχθούν. Κύριε Μπούση, δείχνει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Μπούση. Θα ήθελα να αρχίσω με τα συγχαρητήριά μου επί τη επανεκλογή σα ω Πρόεδρο τη Επιτροπή μα και επίση θα πρέπει να σα ευχηθώ κάθε, κάθε, κάθε επιτυχία. Και εμεί θα συνεργαστούμε ω ΕΛΚ ε, ακόμη καλύτερα μέσα από του υπερδόντε και τώρα έχουμε του ε, αντιπρόεδρου και για τον πρώτο. Την φίλη και συνάδελφο Κίνγκ Γκάλ. Mr. Busutil and for the nomination of Mrs. Kingigal. Any other nominations? Busutil Yagal, έτερος. Thank you, Chair, and congratulations to you. Thank you. Uh, our group... The... Ευχαριστώ, κύριε Χέντα. Εμείς οι σοσιαλιστές θα ψηφίσουμε την ε, κίνηση του Πρόεδρου. There it goes. Second nomination for Mrs. Guns. Δεύτερο ψηφοδέλτιο για την κυρία Γκότς. Και τώρα. Έχει το λόγο κύριε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι κύριε Βέμπερ. Ελπίζουμε να υπάρχει ε, συνεργασία καρποφόρα και κατά το δεύτερο ήμιση. Οι φιλελεύθεροι θέλουμε να προτείνουμε την Σοφία Νετφέλτ ως ε, αντιπρόεδρο τη Επιτροπής μα. Ευχαριστώ κύριε Βέμπερ, κύριε Πρόεδρος. Έχουμε και μία τρίτη. Κύριε Ενέτφελτ, κύριος Μπουσούτη και πάλι. Κύριε Πρόεδρε, για τον τρίτο αντιπρόεδρο θέλω να προτείνω δεν ξέρω αν η κυρία Γκρανίτα Βέμπερ έχει υποψηφιότητα για την πρώτη την Προεδρία, αλλά εμείς για την τρίτη θέση, για τον τρίτο Αντιπρόεδρο μάλλον, θέλουμε να προτείνουμε τον Σαλτορία κολλήνα. Okay. Okay. Then, according to the rules of the... Μάλιστα. Συμφώνως με τον κανονισμό, τα πράγματα θα εξελιχθούν ως εξής. Πρώτον, κύριε Αγκάλ, που σφιόταν. Δεύτερος, κύριε Νετφέλτ. Τρίτος, Για Γιακολίδο και τέταρτος κύριε Γκιόντσα. Συμφωνείτε? Εάν συμφωνείτε με αυτήν την σειρά για τις υποψηφιότητες, ναι. Έτσι έχει πρόταση. Οπότε για να το εκεί είναι οι οποίοι τώρα α, έχουν προταθεί πρέπει να αποδεχθούν και κατόπιν μπορούμε να προχωρήσουμε. Μπορούμε πρέπει να το ρωτούμε, το ζητούμε πρώτα. Εάν ε, υπάρχει κάποια ένσταση να αφορά την ε, ε του, τους, όχι, συνενούν. Συμφωνείτε όλοι. Οπότε και θα σα ψηφίσουμε διαβοήση, Ναι, θεωρούμε ότι έχετε ψηφίσει διαβοή, Κύριε Μπορκέτσιο, ορίστε. Μπορκέτσιο. Απλώς ήθελα να δώσω την αποχή μου. Αποχή λοιπόν και έτσι φαίνεται ότι υπήρξε ε, εκλογή διαβοής. Συγχαρητήρια λοιπόν στους τέσσερις υποψηφίους που μόλις είχαμε. Και μιας και συστήσαμε σε σώμα την Επιτροπή μας. Εκλέξαμε και τα μέλη του ως αντιπρόεδρους. Αν δεν έχετε κάτι στα διάφορα, θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι η ημερομηνία της επόμενης συνεδρίασης έχει οριστεί για την 25η Ιανουαρίου, 9 το πρωί, μέχρι τις 12.30. Και 3 το απόγευμα μέχρι 6.30 το απόγευμα και στις 26 από τις 9 μέχρι τις 12.30. Αυτά λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ.